La seduta è η συνεδρίαση. Έχω μοιραστεί τα κείμενα. Έχετε παρατηρήσει. Please, the floor. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρεμβαίνω για το σημείο 6 των πρακτικών. Δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες επικυρώσαμε την έκθεση που αφορούσε την σύνδεση με την Ουκρανία. Όπως αποτυπώνει μερικώς και το κείμενο των πρακτικών, υπάρχει κάτι το πρωτοφανές εδώ, που είναι η παρέμβαση, η απευθείας μιας πολιτικής προσωπικότητας από το εξωτερικό, από ξένο κοινοβούλιο, μια πίεση έντονη η οποία ασκήθηκε στη συνέλευσή μας και νομίζω ότι αυτό ζημίωσε τη συνένεση που έδωσε το Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση αυτής της έκθεσης. Ακριβώς για αυτό το λόγο σας παρακαλώ να ψηφίσουμε αυτά τα πρακτικά, ούτως ώστε να δούμε αν κάποιοι από τους συναδέλφους, όπως εγώ νομίζω, συμμερίζονται ή όχι αυτή την άποψη που σας εξέφρασα. Και δεν δέχονται την υιοθέτηση λοιπόν των πρακτικών εξαιτία αυτού του πράγματο, λόγω του ότι ε, υπάρχουν προβλήματα σε διαδικαστικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας. Κύριε πρόεδρο, ευχαριστώ. Για να συμπληρώσω αυτά που είπε ο συναδελφός μου. Μία ξένη δύναμη παρενεύει στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή υπάρχει ουσιαστικά μία θέληση να επηρεαστεί η ψήφος των Ευρωπαίων βουλευτών στα πλαίσια της οικονομικής συμφωνίας με την Ουκρανία. Επομένως, αμφισβητούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και θα θέλαμε να ψηφιστούν τα πρακτικά σήμερα για να δούμε αν δεχόμαστε αυτή την ξένη παρέμβαση. Ευχαριστώ. Ε, Κοιτάξτε κύριε Βουλευτά, όχι δεν υπήρχε καμία ξένη παρέμβαση. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Σας άκουσα, άκουσα τις παρεμβάσεις σας. Σας παρακαλώ, ακούστε και εσείς εμένα κανένας δεν υποχρέωσε τους ε, ευρωβουλευτές να ψηφίσουν με τον ΑΒ τρόπο. Δηλαδή, το αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι υπήρχαν ευρωβουλευτές που ήταν υπέρ και ήταν η πλειοψηφία και μία μειοψηφία που ήταν κατά. Είμαστε σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό. Κανένα δεν επηρέασε κανένα. Οι ευρωβουλευτέ είναι ελεύθεροι. Και όσα ελεύθερα όντα δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ακούσουν μια άποψη. Δεν μπορεί μια ξένη βουλή, ένα ξένο ευρωκοινοβούλιο να επηρεάσει συλλήβδιν ευρωκοινοβουλιο να επηρεασει συλλήβδη ολου του ε, ευρωβουλευτές. Έχετε το λόγο, κυρία μου. E, e, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πριν ε, ψηφίσουμε ε, κατά τη διάρκεια της ε, Συνόδου της Ολομέλειας, ψηφίστηκε και το θέμα της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης της Επιτροπής ΑΦΕΤ και εκεί ε, αποφασίσαμε να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία η πλειοψηφία υπέρ ήταν τεράστια και πρέπει να σας πω ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήμασταν ούτε σε τηλεδιάσκεψη ούτε σε απευθείας ε, μετάδοση με άλλο ε, κοινοβούλιο οπότε ήταν μια κυρίαρχη απόφαση που έλαβε η δική μας επιτροπή άρα και το κοινοβούλιο Ευχαριστώ πολύ. Για να συμπληρώσω τα όσα είπε η συνάδελφος, αυτό το οποίο καταγγείλουμε είναι αυτή η παρέμβαση, η απευθείας σύνδεση, η οποία μας παρουσιάστηκε ως ε, συμφωνημένη πράξη, ενώ προηγουμένως δεν είχε συζητηθεί. Και αυτό κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που κάνουν στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Θα έπρεπε λοιπόν η απόφαση να συνδεθούμε απευθεία με την Ουκρανική Βουλή να έχει συζητηθεί και ψηφιστεί. Euh, Κύριε Ευρωβουλευτά, δεν νομίζω ότι οτιδήποτε είναι κατά του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία θα ενισχύσει τους δεσμούς ανάμεσα στα δύο κοινοβούλια, το δικό μας και της Ουκρανίας και νομίζω ότι η ψηφορία του Ουκρανικού Κοινοβουλίου δεν επέβαλε τίποτα σε εμά στους ευρωβουλευτές. Μιλάμε για ελευθερία, για δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι μέλος της ε, Επιτροπής ΑΦΕΤ και η συνάδελφος ε, αναφέρθηκε στην ψηφοφορία εκεί και πρέπει να σας πω πως όπως και, σας, όπως και χτες ανέφερα ε, δεν δόθηκε καν η δυνατότητα στην Επιτροπή ήταν να επανέλθει με οικονομικής φύσης επιχειρήματα για τις συνέπειες τις εμπορικές που θα έχει η συμφωνία αυτή. Η συνεδρίαση στην ΑΦΕΤ έληξε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε δεν νομίζω ότι ακολουθήθηκε η σωστή ε, κοινοβουλευτική διαδικασία ούτε στην Ολομέλεια ούτε όμως και στην διαδικασία της συζήτησης κατά ε, τη διάρκεια της συνάντησης Επιτροπής ΑΦΕΤ. Άρα λοιπόν πιστεύω πως θα πρέπει να διδαχθούμε από τα όσα συνέβησαν, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δεν είστε καν υποχρεωμένος να με ακούσετε. Thank you uh, very much. Uh, I think this is a free, vote. Ε, πρόκειται για κατασυνείδηση ψηφοφορία η οποία διεξήχθη χθες και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε σήμερα τα όσα ψηφίστηκαν χθες. Καταλαβαίνω βέβαια ότι η δική σας θέση είναι διαφορετική, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να αλλάξουμε κάτι. Η Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφασίσει. Οπότε μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε για τα πρακτικά. Η πρότασή σας ποια είναι, συνάδελφε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν για να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε στα χέρια σας. Μπορούμε να ψηφίσουμε διανατάσσεως της χειρός ή με ονομαστική ψηφοφορία. Θέλετε να αλλάξουμε κάτι στα πρακτικά, κάποια λέξη, κάποια φράση. Αυτό ρωτάω θα ήθελα, είναι η απάντηση, να ψηφίσουμε τα πρακτικά για να δούμε αν τα υιοθετούμε και αν δεν τα υιοθετούμε, επειδή δημιουργείται ένα προηγούμενο εξόχως ανησυχητικό, που θα μπορούσε να μας δημιουργήσει προβλήματα με τους εταίρους μας, τα άλλα κοινοβούλια, ε, μπορεί να δημιουργεί ε, ψυχολογική πίεση κάθε φορά που έχουμε τέτοια θέματα. Κατάλαβα, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος είναι κατά της πρότασης αυτής του συναδέλφου, κύριε Γκόμες. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της έγκρισης των πρακτικών Έχετε το λόγο, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η στιγμή. Κρίσιμη, κανονικά. Όταν θέλουμε να υιοθετούμε διεθνείς ή και πολυμερείς συμφωνίες, τα πρακτικά είναι μια σημαντική απόδειξη αυτών. Και τα ψηφίσαμε, ψηφίσαμε αυτή τη συμφωνία σχεδόν με άδεια αίθουσα. ίσως είναι σημαντική αυτή η ψηφοφορία για να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον με αυτή τη συμφωνία. Αντίθετα από αυτά που λένε οι συναδελφοί μου, εγώ νομίζω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να στιγματίσει την νομοθετική μας διαδικασία. Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές, εχθές έγινε εδώ ψηφοφορία και που είναι η έκφραση της βούλησης σημαντικού, σημαντικού τμήματος του Ευρωκοινοβουλίου. Εγώ καταψήφισα εκείνη τη συνθήκη εμπορίου με την, Ουκρανία. Αλλά κανείς δεν μας ανάγκασε. Και ψηφίζοντας υπέρ ή κατά, κανείς δεν υπέστη κάποια πίεση. Η πολιτική αυτή πράξη που εκφράζεται μέσα από την ψηφοφορία αυτή είναι χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες σε σχέση με τα πρακτικά. Το ότι ε, θα μπορούσε να υπονομευθεί αυτή η διαδικασία. Πρόκειται για δύο πράγματα τελείως διαφορετικά. Η πολιτική πράξη επί της ουσίας που ήταν η ψήφιση με το αποτέλεσμα που είχαμε και η έγκριση των πρακτικών ε, ε, είναι ακριβώς η σαφής αντανάκλαση αυτού του γεγονότος. Είναι επικίνδυνο να κάνουμε κάτι άλλο. E Επομένως δεν ε, συζητούμε πια το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Απλώς τη διατύπωση συζητάμε. Όχι το ουσιαστικό περιεχόμενο. Μπορούμε σε τυπικό επίπεδο να προσθέσουμε κάτι, αλλά δεν συζητάμε, δεν αμφισβητούμε το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Επομένω, αυτό που εγκρίθηκε χθε παραμένει εγκεκριμένο. Αυτό είναι τελεσίδικο. Μιλάμε μόνο για κάποιε φράσει που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα πρακτικά. Αλλά δεν αλλάζει το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία και δεν αλλάζει η νομιμότητα της ψηφοφορία. Ήταν απόλυτα νόμιμη αυτή η ψηφοφορία και η σύνδεση με το Κοινοβούλιο του Κιέβου, που δεν επηρέασε την ελευθερία μας. Κανένας Ευρωβουλευτής δεν πιστεύω ότι θεώρησε τον εαυτό του πιεσμένο από οποιονδήποτε. Μόνο η συνείδηση του τον ελέγχει. Όλους μας μας ελέγχει. Τέλο πάντων θα τα ξαναδούμε αυτά και σε νομικό επίπεδο. Παραπέμπω αυτό το σημείο σε μια συζήτηση αργότερα και θα δώσουμε και τεχνικές ε, εξηγήσει. Και πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η δήλωση τη της Κομισιόν και του Συμβουλίου για την αντίρρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακού, ακούστε. Είπα ότι θα στείλουμε αυτή τη θέση που έχει προκύψει για να την ελέγξουμε στο κατάλληλο επίπεδο. Σας παρακαλώ, σταματήστε. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι ξεκάθαρο. Αυτό που έδωσε χθε η ψηφοφορία δεν αλλάζει. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μιλάμε για τη δήλωση της Κομισιόν και του Συμβουλίου για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έξαρση της επιδημίας έμπολα. Εξ του Συμβουλίου. Ο Ιταλός Υπουργός. Presidente. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κύριε Επίτροπε. Η πρόσφατη επιδημία του